Okay, so I'm going to start the meeting and, uh... Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλούμε τους φωτογράφους να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Okay, so we are going to start this extraordinary meeting. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν την έκτακτη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, και θα ήθελα να καλωσορίσω όλους σας. Ε, θα ήθελα να σας καλέσω να βάλετε τα ακουστικά σας, γιατί τώρα θα μιλήσω γαλλικά, τουλάχιστον για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Χαίρομαι που σε υποδέχομαι, Γκρέτα Τιμπέρκ, σε αυτή την συνάθρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Σασόλη ήρθατε τον Απρίλιο του 2019 εδώ και καμιά δεκαριά μήνες μας στείλατε ένα μήνυμα που φαντάζομαι ότι θα μας πείτε ότι δεν κάναμε αρκετά και έχετε προφανώς δίκιο. Θα ξεκινήσω με μια παράθεση. Η κρίση του κλίματος απειλεί την επιβίωση της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε την υπόθεση των καταστροφικών συνέπειων που θα εξαφάνιζαν την ανθρώπινη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Είναι μια παράθεση της Γκρέτα Τούνμπεργκ θα φαντάζεστε. Αλλά δεν το είπε η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Αλλά οι οικονομολόγοι της τράπεζας JP Morgan το είχαν πει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα είναι γεγονότα ανεξάρτητα από εκείνους που τα εκθέτουν και τα παρουσιάζουν και τα αποκαλύπτουν. Και κάποιοι από εσά την αίθουσα αγαπάτε την Γκρέτα Τούρμπεργκ, την λατρεύετε, κάποιοι από εσά την μισείτε, την Γκρέτα Τούρμπεργκ. Όμως τα πραγματικά γεγονότα παραμένουν γεγονότα, επιστήμη επιστήμη και χάνουμε τη μάχη του κλίματος. Εάν σήμερα υποδεχόμαστε και δεχτήκατε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, να σας υποδεχτούμε, κατά την άποψή μου δεν είναι αποκλειστικά για να παίξετε το ρόλο εκείνου που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά για να δημιουργηθούν λύσεις. Διότι δικό σας ρόλος που τον παίζετε με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο είναι να κρούσετε τον κόδωνα του κινδύνου. Και το κάνετε αυτό εδώ και μήνες και μήνες και συναντάτε Συναντήσατε, πιστεύω, εκατοντάδες πολιτικούς υπευθύνου που φωτογραφίζονται μαζί σας, σας λένε αυτά που λέτε είναι υπέροχα και δεν άλλαξαν τίποτα όμως. Και αυτό δεν είναι η νοοτροπία μέσα στην οποία κινούμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε το πνεύμα της Ευρώπης σήμερα και ακόμα λιγότερο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δικός μας ρόλος όταν ακούμε το συναγερμό, είτε προέρχεται από εσά, είτε από του ε, τραπεζικού τη JP Morgan ή του ε, διάφορου επιστήμονε. Ο ρόλο μα είναι να βρούμε λύσει δίκαιε, κοινωνικά, εδαφικά και αξιόπιστες λύσεις, αξιόπιστες επιστημονικά, αξιόπιστες οικονομικά, αξιόπιστες βιομηχανικά. Και καθένας θα παίξει το ρόλο του. Χρειαζόμαστε, και το πιστεύω αυτό, εκ βάθους καρδίας, χρειαζόμαστε την ενέργεια της νεολαίας Καμία κοινωνία δεν μεταμορφώνεται, καμία κοινωνία δεν μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις μας για το κλίμα αν δεν ακούμε ε, την νεολαία μας και δεν παίρνουμε ενέργεια από την νεολαία μας. Και η νεολαία μας σήμερα την εσαρκώνετε εσείς και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μην ξεγελιάσετε Γκρέτα Τούνμπερκ. Σήμερα είσαστε μπροστά σε μια επιτροπή περιβάλλοντος που είναι στην αιχμή, στην πρώτη γραμμή της μάχης για το κλίμα. Δεν είσαστε στο λευκό οίκο με τον Ντόναλτ Τραμπ, ούτε στην Αυστραλία, με έναν πρωθυπουργό που είναι σκεπτικιστή, ούτε με τον Μπολσονάρο στη Βραζιλία, σας στην Ευρώπη, που κάνει την πράσινη συμφωνία και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενέργεια, η ενέργεια της νεολαίας, μια ενέργεια θετική, μια ενέργεια που οδηγεί την κοινωνία, που οδηγεί εκείνους που θέλουν να κινηθούν και εκείνους ε, που είναι πιο διστακτικοί να κινηθούν και αυτό είναι ο δικός μας ρόλος. Λοιπόν, με λίγα λόγια εν είδη Ήθελα να σας συστήσω και σας δίνω το λόγο, ούτως ώστε για 10 λεπτά περίπου να μας μιλήσετε και μετά... Μετά λοιπόν ε, θα έχουμε τη, τους συντονιστές από κάθε πολιτική ομάδα που θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και βεβαίως τους παρακαλώ να τηρήσουν το χρόνο που έχει προεβλεφθεί για κάθε ένα από αυτούς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Hi. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Γκρέτα Τούμπερκ. Εγώ είμαι ακτιβίστρια για θέματα κλιματικής αλλαγής και για τις μελλοντικές εξελίξεις. Για πάνω από 1,5 χρόνο έχουμε θυσιάσει την εκπαίδευσή μας για να διαπαρτηρηθούμε για τη δική σας την αδράνεια. Το Σεπτέμβρη πάνω από 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας από εσάς να ενωθείτε και να στηρίξετε τους επιστήμονες έτσι ώστε να μας δώσετε εν είδη παρακαταθήκης ένα ασφαλές μέλλον. Κατόπιν το Νοέμβρη του 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ανακήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κλιματικής αλλαγής. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι στην αιχμή του δόρατος για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Και αυτό ήταν μια θαυμάσια είδηση. Όταν ε, τα παιδιά σας ε, ή οποτεδήποτε τα παιδιά σας ε, λένε ότι έχει πυρκαγιά, βγαίνετε έξω και μυρίζετε τον καπνό και μετά λέτε ναι πράγματι και εγώ ή καίγεται το σπίτι δεν ήταν λάθος συναγερμός. Όμως ανταυτού εσείς ε, στην περίπτωση που προανέφερα τι κάνατε μπήκατε μέσα, τελειώσατε το δείπνο σας ε, και πήγατε να κοιμηθείτε χωρίς καν να καλέσετε την πυροσβεστική. Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά αυτό δεν βγάζει νόημα. Όταν καίγεται το σπίτι σου δεν περιμένεις ε, λίγα χρόνια ακόμα για να σβήσεις τη φωτιά. Και όμως, παρόλα αυτά, αυτό προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει ε, για την νομοθεσία για κλιματική αλλαγή ε, και τους στόχους μέχρι το 2050 για τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αυτό κατ' ουσίαν σημαίνει ότι παρετήστε. Παρετήστε από τη Συμφωνία των Παρισίων, εγκαταλείπετε τις υποσχέσεις σας και δεν κάνετε ό,τι θα έπρεπε για να διασφαλίσετε ένα ασφαλές μέλλον για τα ίδια τα δικά σας τα παιδιά. Γιατί αυτή η νομοθεσία βασίζεται σε ανεπαρκή κονδύλια, δεν αρκεί ο προπολογισμό για την αντιμετώπιση του διοξιδίου του άνθρακα και ω εκ τούτου έχουμε κάτω από 50% δυνατότητε για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση τη θερμοκρασία στον πλανήτη κατά πάνω από 1,5, ε, από 1,5 βαθμού. Ε, Δυστυχώς ε, δεν ε, χρησιμοποιείται η επιστήμη, δεν αξιολογείται, ούτε τελικά επιτυγχάνονται οι στόχοι της ετήσιας μείωσης της εκπομπής των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η νομοθεσία που προβλέπεται εκπέμπει το μήνυμα ότι πρέπει να λάβουν χώρα ουσιαστικές δράσεις, πράγμα που δεν συμβαίνει. Η αμήλικτη αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συνειδητοποίηση, ούτε σωστή πολιτική. Εξακολουθούμε να βιώνουμε κρίση, η οποία όμως δυστυχώς ποτέ και δεν αντιμετωπίστηκε ως κρίση. Έχουμε πάρα πολλές εξαιρετικές λύσεις, έχουμε ε, μοναδικό πλούτο, κεφάλαια, έχουμε καλή θέληση και πάρα πολλούς ανθρώπους που επιθυμούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν. Εκείνο όμως που δεν έχουμε είναι ευαισθητοποίηση, καθοδήγηση, ηγετικό πνεύμα και πάνω απ' όλα χρόνο. Οι προπολογισμοί για την αντιμετώπιση του προβλήματος του άνθρακα περιορίζονται όλο και περισσότερο και αυτό δείχνει ότι όσο και εάν υπάρχει πρόβλημα, εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτό στη ρίζα του, τότε ε, δυστυχώς ε, θα υπάρξει μόλυνση, ρήπανση της ατμόσφαιρας και ε, πρέπει να εξευρεθεί ένας χάρτης πορείας για να βρεθούν και λύσεις για την ανθρωπότητα. Το περιεχόμενο των κονδυλίων που διατίθενται ή που είναι απαραίτητα δεν ελήφθησαν ποτέ υπόψη στην καθημερινή πολιτική. Ποτέ δεν έγινε λόγο ε, για τα κονδύλια αυτά στα κύρια μέσα ενημέρωση και εσεί τι κάνετε εδώ, προσπαθείτε να χαράξετε πολιτικέ, να συντάξετε νόμου, αγνοείτε όμω ε, την πραγματικότητα και προσπίστε ότι τα προγράμματά σα, η πολιτική σα, αγνώντας τα μηνύματα, κατά κάποιον τρόπο η πολιτική σα, παρόλα αυτά ε, θα αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη κρίση που έπληξε ποτέ την ανθρώπινη ανθρωπότητα. Ένας νόμος ε, ε, που κανείς όμως δεν τον ακολουθήσει, υποτίθεται ότι παρόλα αυτά είναι νόμος. Και γι' αυτό εξακολουθείτε να ε, επιδοτείτε νέες υποδομές που έχουν σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Προσποιήστε ότι το να αγνοήσει κανείς ε, την κλιματική δικαιοσύνη, την ισότητα, αυτό δεν θα θέσει σε κίνδυνο την κατάρρευση της Συμφωνίας των Παρισίων. Προσποιήστε ότι τα κενά λόγια αυτήν την έκτακτη ανάγκη κάπως θα την κάνουν να εξαφανιστεί από μόνη της. Αυτό όμως πρέπει να σταματήσει. Κανένα ε, πρόγραμμα, καμία πολιτική, καμία συμφωνία δεν θα αρκεί όσο συνεχίσετε να αγνοείτε τα κονδύλια που είναι απαραίτητα σήμερα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν χρειαζόμαστε νόμους για το 30 και το 50, χρειαζόμαστε νόμους για το 2020, για φέτος και για κάθε επόμενη χρονιά. Πρέπει να αρχίσουμε να περιορίζουμε ριζικά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην πηγή τώρα αυτή τη στιγμή. Οι απότεροι στόχοι, τι νόημα εάν συνεχιστούν οι ίδιες υψηλέ εκπομπές όπως συμβαίνει σήμερα, αν συνεχιστεί η διακατάσταση και για τα επόμενα χρόνια. Αν συμβεί αυτό, θα δαπανηθούν, θα εξανεμιστούν όλα τα κονδύλια πριν καν έχετε την ευκαιρία να επιδιώξετε έστω την επίτευξη των στόχων του 30 και του 50. Και επειδή λοιπόν αυτές οι τεχνολογίες αρνητικών εκπομπών ε, στις οποίες ε, βασίζεται η επικείμενη νομοθεσία, αυτές οι τεχνολογίες δεν υπάρχουν και δεν ξέρουμε πότε θα υπάρξουν. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, να αλλάξουμε την κοινωνία. Και αυτή είναι μια δυσάρεστη αλήθεια από την οποία δεν μπορείτε να ξεφύγετε όσο και αν το επιθυμείτε διακαώς και όσο σκληρά και αν προσπαθείτε. Και όσο λοιπόν συνεχίζετε να αρνείστε την αλήθεια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η προδοσία που διαπράτετε έναντι των ίδιων των παιδιών σας. Η Ευρώπη πρέπει να καθοδηγήσει. Έχετε αυτή την ηθική υποχρέωση και έχετε μία μοναδική οικονομική και πολιτική ευκαιρία να γίνετε πραγματικά ηγέτες στην αιχμή του δόρατος για την κλιματική αλλαγή. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη για θέματα κλιματικής αλλαγής. Εσείς το είπατε ότι αυτή η απειλή είναι υπαρξιακή. Ε, τώρα έχει έρθει η στιγμή να αποδείξετε ότι εννοείται αυτά τα οποία λέτε. Και εμείς δεν θα ικανοποιηθούμε με τίποτα λιγότερο από αυτά που λέει η επιστήμη και από αυτά που μας δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να διαφυλάξουμε τις συνθήκες διαβίωσης, όπω όπως τις γνωρίζουμε και για το μέλλον. Οτιδήποτε άλλο σημαίνει παρέτηση. Αυτή η νομοθεσία για το κλίμα είναι παρέτηση γιατί η φύση δεν διαπραγματεύεται και δεν μπορεί κανείς ε, να συνάψει συμφωνίες και νόμους με φυσικά φαινόμενα. Εμείς λοιπόν δεν θα σας επιτρέψουμε να ε, παρετηθείτε και να μας εγκαταλείψετε στο θέμα του μέλλοντός μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται από τους συντονιστές τους στην ΕΝΒΗ. Από το ΕΛΚ ξεκινάμε. Πίτερ Λίζε, για έξι λεπτά. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Γκρέτα. Πολύ εντυπωσιακή η δήλωσή σου. Και ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειες που κάνεις τους τελευταίους μήνες. Για μένα είναι σημαντικό που εκπροσωπεί σε εκατομμύρια νέους ανθρώπους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Συναντώ στην εκλογική μου περιφέρεια πολύ συχνά εκπροσώπους της, του κινήματός σου και εντυπωσιάζομαι πόσα πράγματα ξέρουν και πόσο ε, αφοσιωμένοι είναι στο έργο τους. Συνάντησα μία νέα κοπέλα που ταξίδεψε ε, σε μια εκδήλωση Παρασκευέ για το μέλλον, 25 χιλιόμετρα μόνο, αλλά χρειάστηκε τρει ώρε. Γιατί δεν ήθελε να ζητήσει να την πάει κάποιο με αυτοκίνητο, χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζική μαζικής ε, μεταφορά και ε, πολλά τέτοια παραδείγματα συνάντησα. Η επιστημονική προσέγγιση είναι σαφή. Όταν όλα τα μέρη συμφώνησαν να βάλουν κάποια μέτρα και συμφώνησαν ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από τρει βαθμούς και διατρέχουμε τον κίνδυνο να περάσουμε το σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως όταν λιώσουν οι πάγοι της Γρυλανδίας ή όταν λιώσουν και οι παγετώνες του βορείου ημισφαιρίου. Καταλαβαίνω τι κίνητρο έχει νέα γενιά. Τα παιδιά μου είναι μόλις λίγα χρόνια πιο μεγάλα από σένα. Αν δεν δράσουμε σύντομα, θα έχουμε την κατάσταση ίσως σε 30-40 χρόνια όπου η νέα γενιά και τα παιδιά σου δεν θα είναι σε θέση να ελέγξουν τις αλλαγές του κλίματος πλέον. Γι' αυτό όλα τα μέρη, όλα τα κόμματα πρέπει να κάνουν περισσότερα από αυτά που δεσμεύτηκαν να κάνουν στη Συμφωνία των Παρισίων. Όλα τα συμβαλόμενα μέρη της Συμφωνίας θα κάνουν περισσότερα για την πολιτική μου ομάδα, το ΕΛΚ. Θα τόνιζα τρία συγκεκριμένα σημεία τα οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε. Πρώτα απ' όλα Θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και στην καινοτομία, παραδείγματο χάρη, για να μειωθεί η χρήση άνθρακος από τη βιομηχανία. Πρέπει να είναι εφικτό, πιστεύω. Είναι δυνατόν η βιομηχανία να παραμείνει, αλλά να γίνει πιο καθαρή και πιο φιλική προς το κλίμα. Και έτσι να δείξουμε το δρόμο και σε άλλε μεγάλες οικονομίες, όπω είναι η Κίνα, όπω είναι η Ινδία. Και είναι τεράστια προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε ενωμένοι. Το πρόβλημα είναι τα κράτη-μέλη, Υπουργοί Οικονομικών και Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων που προτείνουν περικοπέ όσον αφορά τα κονδύλια για την καινοτομία και γι' αυτό πιστεύω ότι εμείς όλοι πρέπει να πολεμήσουμε ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να δεχθούν τις ε, ευθύνε τους. Δεύτερο σημείο, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα ευρωπαϊκά δάση. Λόγω της αλλαγής του κλίματος έχουμε ξηρασία, έχουμε κύματα καύσωνος τα τελευταία χρόνια και τα ε, επιχειρήσεις ε, έχουν πρόβλημα όσον αφορά την εκμετάλλευση των δασών. Είναι πολύ σημαντικά τα δάση για το κλίμα, το σημαντικότερο στοιχείο που έχουμε στην Ευρώπη και ένα καλό παράδειγμα που δείχνει ότι τα οικονομικά και τα κλιματολογικά προβλήματα πάνε χέρι με χέρι ε, και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τρίτον, είμαι αποφασισμένο, πολύ αποφασισμένο πάνω σε αυτό. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή ε, ε, κτιμή για τον άνθρακα και σε περιοχές που δεν υπάρχει, στις μεταφορές και στα κτίρια. Και για να φτάσουμε εκεί, μπορούμε να φτάσουμε για τον φόρο ε, και είναι ομόφωνη απόφαση με όλα τα κράτη-μέλη που χρειάζεται και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε όσον αφορά το φόρο άνθρακα και γι' αυτό και για, αυτούς, και διάφορους τομείς υποστηρίζω το ETS το εμπόριο ε, εκπομπών άνθρακα. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό να έχουμε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα χωρίς να μην έχουμε μια προσέγγιση για την τιμολόγηση για το κόστος του άνθρακα στην Ευρώπη. Λοιπόν, κατάλαβα το μήνυμά σας όσον αφορά το κλίμα, αλλά πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι η νομοθεσία για το κλίμα που θεσπίσαμε είναι φιλοδοξή για να φτάσουμε σε δετερότητα για τον άνθρακα. Είναι φιλόδοξη αυτή η πολιτική για να πετύχουμε τους στόχους του 2030 ακόμα και αν πάμε από 40 μέχρι 50% είναι σημαντικό βήμα. Ποια είναι η ησυχία μου. Δεν ξέρω καμία άλλη μεγάλη οικονομία στην Ιφίλιο που να εξετάζει τέτοια ενδεχόμενα και το να κάνει τέτοιο βήμα. Και αυτό είναι το τελευταίο μου βήμα. Ε, πέρασε στον Ατλαντικό. Συνάντησες πάρα πολλούς ανθρώπους στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στη Λατινική Αμερική και θα ήθελα να καταλάβω τι έμαθες. Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητα σε αυτές τις χώρες, να τις κινητοποιήσουμε και άλλους όπως Κίνα, Νότια, Αφρική, Ινδία, Ιαπωνία να αυξήσουν τους στόχους τους. Μίλησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χτες και δεν υπάρχει άλλη μεγάλη οικονομία, μόνο μικρές χώρες που θαυμάζω πάρα πολύ, το Μαρόκο, η Κωνσταντίνα, η Αιθιοπία, αλλά δεν αλλάζει ε, η σημαντική ποσότητα των εκπομπών. Αυτοί που παράγουν τι περισσότερε εκπομπέ και θα πρέπει να γυθούμε μέσω παραδείγματο. Αυτή είναι μια πολύ σαφή απάντηση, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί. Λοιπόν, πώς μπορούμε να πείσουμε άλλες μεγάλες οικονομίες στη Λατινική Αμερική και σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι αυτό που πιστεύω ότι είναι σαφέστατο από επιστημονική πλευρά είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στην κυρία Γκούτελαντ, συντονίστρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και εισηγήτρια για τον κλιματικό νόμο. Για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα, Γκρέτα. Θα μιλήσω σου Είναι τιμή μας που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μας και είναι χαρά μου να μιλώ σου ειδικά στην αίθουσα και να με καταλαβαίνεις απευθείας. Βεβαίως, θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές και θέλουμε οι φωνές υπέρ του περιβάλλοντος να υψωθούν ε, ε, ακόμα πιο ε, ηχηρές. Και αυτό αισθάνθηκα όταν ε, πήρες εδώ το λόγο και άρχισες να μιλάς. Ε, σε ευχαριστούμε για τη σκληρή σου δουλειά, για σένα και για όλη τη γενιά που εκπροσωπείς. Είμαι μέλος του Ευρωκοινοβουλίου εδώ και έξι χρόνια. Και βλέπω το πριν και το μετά ε, σε σχέση με τις παρασκευές για το κλίμα, για το μέλλον, το Fridays for Future. Έχεις δίκιο λοιπόν, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Συζητούμε τα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών, όχι μόνο τον κλιματικό νόμο που σήμερα υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ είμαι συγγήτρια για το νομοθέτημα αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο η Ευρώπη έχει και την ευθύνη αλλά και τις δυνατότητες, τους πόρους για να ε, πραγματοποιήσει μια δίκαιη μετάβαση. Πρέπει όλοι να βεβαιωθούμε ότι αυτό γίνεται, αλλά η μετάβαση να είναι σαφώς δίκαιη, να καλύπτει όλους τους ε, τομείς και να είναι δίκαιοι και απέναντι σε όλου του πολίτε. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε στου διάφορου μηχανικού τομεί, αλλά και στα διάφορα μέρη του κόσμου, στι διάφορε γεωγραφικέ περιοχέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω έχει μια φωνή με κύρος, η οποία πρέπει να ακουστεί, αλλά έχει και επιπλέον ευθύνε να μειώσει τι εκπομπέ τη ευθύ αμέσω. Το συνειδητοποιούμε αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό να δώσουμε ήδη εμείς ένα καλό παράδειγμα και να επηρεάσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Να φανεί ότι το εννοούμε και ότι μειώνουμε εμείς πρώτοι δραστικά τις εκπομπές μας. Δεν είναι θέμα απλώς δικαιοσύνης, είναι και θέμα φιλοδοξίας. Πρέπει να είμαστε φιλοδοξότεροι και αυτό είναι κάτι που το έχεις πει επανειλημμένος στις ομιλίες σου, όπως και σήμερα. Ο στόχος του να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι στο 2050 είναι ένας στόχος που δεν μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Πρέπει να θέσουμε φιλοδοξότερους στόχους αμέσως ε, και σήμερα και για τα επόμενα χρόνια. Και Όπω λε και εσύ, ο κλιματικό νόμο που προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα δεν συμφωνεί με τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε. Δεν ικανοποιεί ούτε σένα ούτε εμά. Όμω θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι τα πράγματα θα πάνε γρηγορότερα, ότι θα δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία και ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον κόσμο. Εγώ θα δώσω τη δική μου μάχη ω εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Ελπίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι μια δύναμη που θα αγωνιστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα για να συμπαρασύρει ε, σε αυτή τη μάχη. Και ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν πριν τη Γλασκόβη. Ε, να γίνει εδώ το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς και να δώσουμε εκεί πραγματικά ένα καλό παράδειγμα. Ο κλιματικός νόμος πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα με έναν προπολογισμό που να προβλέπει την απαλλαγή από τον άνθρακα μαζί με, ε, με τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει να δούμε πώς προχωρούν αυτά παράλληλα. Θα εργαστούμε πολύ σκληρά, αλλά να είσαι βέβαιη ότι η δική σου δουλειά μας ε, βοηθά, μας εξυπηρετεί με την πίεση που ασκείται στο Κοινοβούλιο και τα επιστημονικά πορίσματα, οι επιστημονικές συμβουλές θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα και ο πύχη βάσει του οποίου θα καθορίζουμε τι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν θέλω όμω και να σε ε, ξεγελάσω, ούτε να πω ότι όλα αυτά θα γίνουν ε, με κάποιο τρόπο απλό. Υπάρχουν πολλέ δυνάμει εδώ στο Κοινοβούλιο και παρατάξει που αντιμάχονται τι ε, αλλαγέ υπέρ του κλίματος. Συντηρητικέ δυνάμεις που θέλουν να αποδυναμώσουν τη δουλειά που κάνουμε. Ελπίζω να το γνωρίζει. Υπάρχει μεγάλο διχασμός στο Ευρωκοινοβούλιο μεταξύ όσων θέλουν να κάνουν κάτι αμέσω και όσων δεν θέλουν. Ε, φαντάζομαι ότι το γνωρίζεις ήδη, αλλά καλό είναι να το πω ξανά εδώ, μπροστά σε όλους, μιας και είμαστε παρόντες στην ίδια αίθουσα. Μιλάμε την ίδια γλώσσα και με καταλαβαίνεις. Περνάμε τώρα σε ένα σημείο καμπή, ένα σημείο όπου θα γίνεται το ένα και πιο δύσκολο να υλοποιήσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων πλήρως. Ε, πρέπει να γίνουν περισσότερα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά η δουλειά για το κλίμα αγγίζει τη ζωή όλων των ανθρώπων. Έχουμε δεσμευτικού στόχου για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για την ενεργειακή απόδοση, για την ε, εμπορία δικαιωμάτων ε, εκπομπών, για τι εκπομπέ από τον τομέα των μεταφορών. Έχουμε πολλέ δυνατότητε ήδη. Είναι μια ευκαιρία για περισσότερε προσπάθειε, νέε προσπάθειε που στοχεύουν σε μια ε, κλιματικά ουδέτερη κοινωνία. Μπορεί μετά τη μετάβαση να έχουμε βελτιώσει αρκετά τα πράγματα και είμαι πεπισμένη ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχο μα. Θέλω λοιπόν να βεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί αυτό. Εμεί ω σοσιαλιστέ και δημοκράτε θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, η ομάδα SND, θα παρακολουθεί διαρκώ τα θέματα ισότητα και δικαιοσύνη, μια δίκαιη μετάβαση, γιατί για μα είναι πρώτε τη σημασία να βεβαιωθούμε ότι η ευημερία, η ασφάλεια και η κλιματική ε, ε προχωρούν χέρι-χέρι. Θέλουμε μια πιο καλά εξισορροπημένη κοινωνία και θέλουμε αυτό να γίνει γρήγορα. Να κλείσω λέγοντα ότι εκπροσωπεί μια γενιά ανθρώπων που μετά την έλευση του νέου αιώνα ε, δίνουν μια μάχη για τον πλανήτη μα, για το κλίμα και το περιβάλλον μα. Ευχαριστώ λοιπόν και εσένα και όλου του νέου ανθρώπου που ακολουθούν τα βήματά σου. Οι πρωτοβουλίε σου και η αλήθεια που φανερώνει στην κοινωνία μα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ε, το ε, παρατηρούμε και το σεβόμαστε και το αξιοποιούμε πλήρως τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ασκούμε πίεση και θα είμαστε αμήλικτοι. Θέλουμε να γίνουν περισσότερα και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ευχαριστούμε που ήρθες. Okay. Let's say that Πολύ ωραία. Σας ε, έδωσα λίγο χρόνο ε, για κάποιο λόγο, επειδή κάνατε και ένα είδος ρεπορτάζ, ας πούμε, Με πάση περιπτώσει, ε, πρέπει να προσέχουμε το χρόνο. Χαίρομαι που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Γκρέτα, καλώς ήρθες και πάλι. Την τελευταία φορά που ήσουν εδώ, πολλοί πολιτικοί ήθελαν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία και όταν οι πολιτικοί ασχολούνται με προεκλογική εκστρατεία υπάσχονται πάρα πολλά και μετά υπαναχωρούν και κάνουν πολύ λιγότερα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν επιτύχαμε έστω κάποια βελτίωση. Στην COP21 είπαμε ότι θα έχουμε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα ε, μέχρι το 2050. Μας λες ότι αυτό δεν αρκεί, αλλά σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Επίσης, ε, ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια αρκετά ε, δύσκολη συζήτηση για το θέμα της κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Πολλοί υπερψήφισαν, αλλά και αρκετοί καταψήφισαν. Υπήρξαν πολλές κριτικές όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Αλλά για ρίξτε μια ματιά στον κόσμο. Δεν σε τι γίνεται. Έχουμε δασοπυρκαγιές, ε, πλημμύρες, ε, πολλά φυσικά φαινόμενα. Γι' αυτό όταν ανακηρύξαμε την κλιματική έκτακτη ανάγκη, ίσως ε, να μην απήχαμε και πολύ από την πραγματικότητα. Αν δείτε τη Βαλτική θάλασσα, εκεί μπορείτε να δείτε πως η Βαλτική επηρεάζεται. Έχουμε πολύ πιο ήπιους ε, χειμώνες, ε, πέφτει η στάθμη της θάλασσας. Αυτά όλα πολύ γρήγορα ε, και αυτά θα επηρεάσουν σαφώς τη βιοπικιλότητα. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω ιδιαίτερα εκ μέρους Κατρίν Σαπό, μιας ευρωβουλευτήνας ε, που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Είναι η πρώτη γυναίκα που με ένα χέρι ε, διέσχισε όλο τον κόσμο με το ιστιοπλοϊκό της. Οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το 50% της αυξημένης ε, θερμοκρασίας στον πλανήτη. Αυτές λοιπόν οι τεράστιες ποσότητες θερμότητας που απορροφούν οι ωκεανοί Αυτές οι τεράστιες ποσότητες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν και χρειάζονται μακροχρόνιες και σκληρές προσπάθειες για να πετύχουμε τους στόχους μας μέχρι το 2050 και μεταγενέστερα. Ε, και εγώ τότε, ξέρετε, θα είμαι ηλικία 105 ετών. Ε, δεν ξέρω από πού θα κοιτάω τη γη, από πάνω ή από κάτω πάρα πολύ πολιτικοί το παίρνουν αυτό πολύ ελαφρά. Ε, ίσως ε, να είδατε κάποιους ε, στο Twitter στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που πιστεύουν ότι με ένα tweet μπορούν να λύσουν τα προβλήματά μας. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι κακό παράδειγμα για όλους μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι καινοτομία. Και όταν μιλάμε για καινοτομία υπάρχουν κάποιες χώρες που τα καταφέρνουν πολύ καλά μπορείτε να δείτε τις καινοτόμες χώρες στην Ευρωπή. Ε, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, αυτές είναι οι χώρες που έχουν ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα και προηγούνται. Βεβαίως εσύ ε, δεν πας σχολείο ε, έχεις εγκαταλείψει το σχολείο σε κάποιο βαθμό. Από την άλλη βέβαια έχουμε ένα πολύ καλό σχολικό σύστημα και Χαίρομαι που ε, ασκεί πολιτική πίεση, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπαμε καμία κινητοποίηση στις Βρυξέλλες. Ε, Ευχαριστώ. Επόμενη ομάδα, η ομάδα ID. Σέλβια Σαρντόνα για τρία λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Γκρέτα. Αυτήν την εβδομάδα το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένη πρόσβαση για τους ε, υπαλλήλους, για συνεργάτες και βουλευτές ακόμα. Όμως είναι ανοιχτό ε, για την Κρέτα. Με εκατοντάδε εδώ ανθρώπου φαίνεται ότι οι οικολόγοι δεν κολλάνε κανέναν ιό. Μην με παρεξηγείτε, εκτιμώ πάρα πολύ του νέου που πιστεύουν σε κάτι όπω η Κρέτα και που με πάθο και αφοσίωση μάχονται για κάποιο ιδανικό. Δυστυχώ όμω είναι τελείω εμφανέ ότι την Κρέτα την, την εκμεταλλεύονται ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα τη και να την κάνει καλύτερα. Όμω, ε, αντιδιαστολή με όσου εδώ τη χειροκροτούν, εγώ δεν θέλω να είμαι ε, υποκρίτρια μπροστά στην Κρέτα. Πιστεύω ότι οι μάχες των ε, ε, οικολόγων, των δίθεν οικολόγων, ε, είναι γεμάτε υποκρισία, λάθη και τιμωρούν τον κανονικό κόσμο. Είναι υποκριτέ, διότι ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά θέλουν μια αποανάπτυξη που θα του οδηγήσει στην ευτυχία. Ποιοι θέλουν να παρατήσουν τα smartphone και το 5G. Ποιοι θέλουν να ε, σταματήσουν να ταξιδεύουν με αεροπλάνα που τα κοστίζουν 19 ε, ευρώ η πτήση. Ποιοι θέλουν να σταματήσουν να πίνουν αναψυκτικά με ζάχαρη και να τρώνε fast food. Ή να πλένουν στο δυνατόν λιγότερο τα ρούχα του ή να βάζουν βάζουν στο maximum, στο full το air condition. Ε, είναι ε, ε, πραγματικά γνωστά όλα αυτά σε όσους προσελτίζονται από τη θρησκεία του, της οικολογίας ε, και τι θέλετε να κάνουμε, να ξαπλώσουμε έναν ιό για να μειωθεί ω το δυνατόν περισσότερο η ρήπανση στην Κίνα, είναι αυτό λύση. Διότι όταν κλείσουν οι εταιρείε λόγω τη ρήπανση θα έχουμε και περισσότερη ανεργία και φτώχεια. Και υπάρχουν και πολλά σφάλματα εδώ, γιατί βλέπουμε ότι η Γκρέτα και οι συμμαχοί τη διοργανώνουν διαδηλώσει και τελετουργίε και συγγνώμη, λιτανίε ε, σε όλο τον κόσμο. Όμω οι οικολόγοι ποτέ δεν αναφέρουν χώρε όπω η Κίνα και η Ινδία, ούτε οργανώνουν ε, διαδηλώσει σε εκείνε τι χώρε. Η Κίνα έχει αυξήσει την κατασκευή εργοστασίων του άνθρακα μέχρι το 2030 και έχει 7 στι 10 πιο μολυσμένε πόλει στον κόσμο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ε, φόροι για το πλαστικό, τα, τη, ζάχαρη, τα καύσιμα και τελικά την πληρώνουν οι απλοί πολίτε. Ε, κατηγορούμε του καταναλωτέ για κλιματική εγκλήματα. Γιατί, γιατί μπορούν να τρώνε κανονικά κάποιες φορές και κρέα, γιατί μπορούν να αγοράσουν κάποτε ένα σπίτι, να πληρώνουν ένα σπίτι και κάποιες φορές και ένα αυτοκίνητο. Πραγματικά ε, ο κίνδυνο είναι οι ιδέες αυτές ε, να τιμωρούν τελικά καταναλωτές και ε, εταιρείε και να δημιουργούν μεγάλες κοινωνικές ζημιέ. Ε, η αποβιομηχανοποίηση πολλές φορές σημαίνει και φτώχεια και θέλουμε να μην γίνουμε δέσμοι μιας υποανάπτυξης, υπανάπτυξης η οποία θα είναι μόνιμη. Ε, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ρήπανση, ε, δεν θέλουμε να το αρνηθούμε. Το αντίθετο όμως χρειάζονται επιστημονικά στοιχεία και όχι ένα λαϊκό δικαστήριο από παρακινητές όπως αυτοί που εκμεταλλεύονται την Κρέτα. Πρέπει να πάψουμε τα ιδεολογικά σλόγγαν με προγράμματα τα οποία είναι ανέφικτα και που τιμωρούν πολύ συχνά αυτούς που δεν φταίνε. Με συγχωρείτε, ε, λίγο σεβασμό στον άλλο, στους άλλους δώσατε 1,5 λεπτό παραπάνω. Ε, δημοκρατία θέλουμε, υποτίθεται να έχουμε εδώ. Ιδάλλως είναι δύσκολο να κοστούν όλες οι απόψεις. Ευχαριστούμε, το πήραμε το μήνυμα. Οι πράσινοι έχουν τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο και θα μ' ακούτε. κ. Έκχοτ. Καταρχά, καλώ ήρθε, Γκέτα Τούμπερκ. Καλώ επανήλθε και καλωσορίζουμε όλου την αίθουσα που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τι πολιτικέ, για το κλίμα που προσπαθούμε να απογειώσουμε εδώ. Ποτέ δεν είδαμε τόσο μεγάλο πλήθο εδώ. σω μπορούμε να κρατήσουμε του αριθμού, γιατί του χρειαζόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε τα θέματα του κλίματο και την κοινομοθεσία. Έχει δίκιο και ευχαριστώ πάρα πολύ που πραγματικά επανέφερε το θέμα τη επιστήμη. Διότι αυτό είναι το κρίσιμο σημείο εδώ πέρα. Κάθε φορά όταν ακούμε ομιλίε από κάθε πολιτικό, που αναφέρονται στη σημασία του κλίματο και την κατεπίκουσα ανάγκη για το κλίμα. Σαν πράσινη πάντα λέγαμε ότι δεν αφορά το θέμα τη λέξη, αλλά τη δράση. Δυστυχώ όμω, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνη να αυξήσει ε, τις προσπάθειες όταν υπέβαλε την πρόταση για την Πράσινη Συμφωνία. Ελπίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πραγματικά θα μετέτρεπε την, ε, το Πράσινο Σύμφωνο σε δράση. Σήμερα παρουσίασαν το νόμο για το κλίμα και είναι άκρος απογοητευτικός φέτος θα έπρεπε να είχε χρονιά που θα φορούσε την αύξηση των φιλοδοξιών μας. Και Πίτερ Λίζε, σωστά τα είπες. Είχες απόλυτο δίκιο. Πρέπει να αυξήσουμε τη φιλοδοξία μας. Και η ερώτησή σου, πώς να το πετύχουμε αυτό, δείχνοντα ότι μπορούμε εμείς να το κάνουμε, ότι το κάνουμε. Αλλά αν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός της νομοθεσίας για το κλίμα λέει ότι θα κάνει μια πρόταση μέχρι το Σεπτέμβριο που ίσως να αυξήσουμε κάτι για τι φιλοδοξίε για τι εκπομπέ το 2030, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Διότι η Συμφωνία των Παρισίων οικοδομήθηκε τόσο ώστε κάθε πέντε χρόνια να έχουμε μία όθηση. Και το 2020 είναι η χρονιά, ο Νοέμβριο του 2020 είναι η στιγμή στη Γλασκόβη που αυτό θα πρέπει να συμβεί. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, ποιο θα είναι έτοιμο. Η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία. Όχι, εάν εμεί δεν είμαστε έτοιμοι. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι ίσως έχουμε πρόταση μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι κάτι που θέτει εν κινδύνο τη Συμφωνία των Παρισίων. Διότι αν δεν αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας και δεν πετύχουμε παγκόσμια όθηση για την, την αύξηση των εκπομπών, επί πέντε χρόνια θα ακολουθούμε την παρούσα πορεία και η παρούσα πορεία ε, μας οδηγεί σε μια αύξηση θερμοκρασίας πάνω από τις βαθμούς. Αυτή είναι η τάση που ακολουθούμε. Και πρέπει τώρα να αλλάξει αυτή η πορεία και η Ευρώπη θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Τώρα, στην νομοθεσία περί κλίματος μπορούμε να έχουμε καλές συζητήσεις στις Βρυξέλλες, στη Φυσαρίδα των Βρυξελών, περί κατεξοδότησης πράξης, περί εκτελεστικών πράξεων, αλλά όλα αυτά υποτίθεται τα μέτρα θα ξεκινήσουν μετά το 2030. Δεν θα πρέπει να το κουβεντιάζουμε αυτό. Η συζήτηση θα έπρεπε να αφορά το τι θα αυξήσουμε, πόσο θα αυξήσουμε τη δράση τώρα και πώς θα δημιουργήσουμε μια όθηση σε όλο τον κόσμο και είναι κάτι που απελπισμένα το χρειάζεται ο κόσμος. Η προθεσμία για τον Νοέμβριο ε, είναι εκεί. Περνάει ο χρόνο, πρέπει να δυστηριοποιηθούμε. Ευχαριστώ, Γκρέτα, που έθεσε στο θέμα τη επιστήμης. Ευχαριστώ και εσά για τα χειροκροτήματα. Αλλά εσεί θα πρέπει να οδηγήσετε και στη δράση, όχι μόνο στα χειροκροτήματα. Thank you Ευχαριστώ το πολύ εκ μέρους του ΙΣΙΑ Πιάτικο Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ε, είχαμε την ε, νομοθεσία για το κλίμα ε, όπου καθορίζονται οι στόχοι για ουδετερότητα μέχρι το 2050. Έχω αρκετές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρηθούν όλοι οι στόχοι μετά το 2030 μέσα ε, από κατεξουσιοδότηση πράξη. Και αυτό είναι ένα πολύ ε, ανεπαρκές νομικό εργαλείο. Επιπλέον, Ακόμα και η πράσινη συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι γεννήθηκε, είναι απολύτως απαραίτητο όλες οι πολιτικές να αξιολογούνται έχοντας κατά κύριο λόγο κατά νου την αύξηση των στόχων του 2030. Το ECR, η ομάδα μας, ε, είναι κατά της ε, αύξησης ε, των ορίων, γιατί θα υπάρχει και νομική ασάπια, όπως έχει επανειλημμένα εκφράσει η προηγούμενη Επιτροπή. Η θέση της πολιτικής μας ομάδας, του ECR, είναι η εξής. Πρώτον, να μην αλλάξουμε τους στόχους να παραμείνουμε προσιλωμένοι στη Συμφωνία των Παρισίων. Ε, δύο, δεύτερον, να υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου από τεχνική, κοινωνικονομική, τεχνική σκοπιά. Ε, θέλουμε καλύτερο προγραμματισμό και λιγότερους συμβολισμούς. Τρίτον, να δημιουργήσουμε ομάδες ποιήσης για να ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο ε, αν δεν υπάρχει γενικότερη παγκόσμια συνεργασία και εδώ υπενήσουμε πάλι την Κίνα και την Ινδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να αλλάξει τίποτα σε θέματα κλίματος και βεβαίως θα καταστραφεί η οικονομία μας. Ε, θέλω να, να ολοκληρώσω με ένα κάπως ε, ασήμωτο τρόπο, αν μου επιτρέπετε, Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Κρέτα για το ότι διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο κοινό για αυτό το θεμαλιό, κεφαλαιόδες θέμα. Επιτρέψτε μου όμως να της δώσω και μία συμβουλή ως πατέρας προς κόρη να πας στο σχολείο. Σχολείο να πας και να αρχίσεις και να κάνεις μία κανονική ζωή. Η παιδική σου ηλικία είναι εξίσου πολύτιμη όπως και το κλίμα. Και αν δεν κάνεις κάτι για την παιδική σου ηλικία θα τη χάσεις για πάντα. Ακριβώς όπως και αν δεν κάνουμε κάτι για το κλίμα θα χάσουμε το παιχνίδι για πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρει περισσότερα για τις επιστήμες από ό,τι πολλοί από εμάς. Μόντικ Κουέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ θα μιλήσω σουηδικά. Είναι η κοινή μας γλώσσα. Γεια σου Γκρέτα, ε, καλώς ήρθες εδώ. Ε, πρώτα απ' όλα για την ομάδα μου. Από την πλευρά όλων μας θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όσα κάνεις από την gue Ευχαριστούμε που δίνεις φωνή σε όλους τους νέους που θέλουν να γίνουν περισσότερα, περισσότερα στην ε, διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων. Ευχαριστώ λοιπόν για τον αγώνα που δίνεις. Διευκολύνεις τη δουλειά μας γιατί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το κλίμα. Βλέπω βεβαίως σήμερα ήδη πολλές ε, εκδηλώσεις ε, υποκρισίας σε αυτή την αίθουσα. Έχουμε πολλά στοιχεία επιστημονικά για το κλίμα. Οι αποφάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν ε, είναι δυνατόν να ληφθούν. Αλλά δεν υπάρχει τόλμη, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις. Ελπίζω η ομιλία σου σήμερα εδώ να έχει τη βαρύτητα που, θα, που της αρμόζει. Βεβαίως, είναι ωραίο να χρησιμοποιήσει ως σύμβολο για τον ακτιβισμό υπέρ του κλίματος, αλλά είναι σημαντική και η άποψη που εκφράζει, η φωνή σου, γιατί κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη. Ε, ο κλιματικός νόμος, οι κλιματικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι αρκετά φιλόδοξες. Μείωση 50% στα 2030 για τις εκπομπές δεν είναι αρκετό. Είναι σαφές αυτό, είναι επιστημονικά τα δεδομένα. Πρέπει να φτάσουμε σε επίπεδο φιλοδοξιών όπως αυτό που μας συστήνουν οι επιστήμονες. Και αν ήμασταν ευφύης, θα, θα αυξάναμε κι άλλο το επίπεδο των στόχων μας για να είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι. Ε, ίσως με συγκέντρια την κυρία Γκούτελαντ να πετύχουμε κάποια πρόοδο και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη θέση του Ευρωκοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι γίνεται και σε άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάναμε στο παρελθόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Θα είμαστε στο πλευρό σου. Σε ευχαριστώ. Okay, the Τελευταίος ομιλητής. Ελεονόρα Εύη, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητή Γκρέτα, χαίρομαι ιδιαίτερο που σε συναντώ εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, μια έκκληση. Βοήθησέ μας να μιλήσουμε για την έλλειψη διαφάνειας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ξέρεις ίσως ότι εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο, εργαζόμαστε με καλό βαθμό διαφάνεια. Οι συζητήσει είναι δημόσιε, στο διαδίκτυο, οι τροπολογίε δημοσιεύονται και μεταφράζονται. Αυτό βοηθά τη δημοκρατία. Επίση, συχνά μα έχει οδηγήσει σε πολύ φιλόδοξε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μα έχει βοηθήσει αυτό, κυρίω όσον αφορά τα θέματα του κλίματο και του περιβάλλοντο κατά παρελθόν. Αντιθέτω, ε, το Συμβούλιο, όπου είναι οι εκπροσώποι των κρατών μελών, είναι μια μαύρη τρύπα δεν υπάρχουν ε, ε, πρακτικά, δεν υπάρχουν καταγραφέ ε, των θέσεων των κρατών μελών για κάθε θέμα και γίνεται κυκλισμένων των θηρών συζήτηση. Δεν ξέρουμε αν επικρατούν τα δημόσια συμφέροντα ή όπω συχνά γίνεται τα εθνικά ή άλλα συμφέροντα επικρατούν. Σου ζητώ να μα βοηθήσει όσον αφορά αυτή τη μάχη και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά αυτή την διαφάνεια. Κλείνοντα η χώρα μου, η Ιταλία, σήμερα έκανα πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση, καθόρισε στη μόνιμη αντιπροσωπεία εδώ στην ένα μητρό διαφάνεια εδώ στι Βρυξέλλε για να καταγράφονται τα διάφορα λόμπι και ομάδε συμφερόντων. αλλά πολλά πρέπει να γίνουν για τη διαφάνεια στο Συμβούλιο και να εξασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε του φιλόδοξου στόχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Ευχαριστώ. Thank you, sir. Unless... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, εάν η Γκρέτα δεν θέλει να ξαναλάβει το λόγο, που δεν νομίζω ότι θέλει, λύεται η συνεδρίαση, κλείνουμε τη συνεδρίασή μας και με την Κρέτα θα πάμε στο πίσω μέρος του αίθουσα. Αφήστε τις λοιπόν λίγο χώρο, αν δεν έχετε αντίρρηση. Και Ελπίζω στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, Περιβάλλοντος ε, που θα συζητηθεί η κλιματική νομοθεσία να είμαστε εξίσου πολλοί όσοι ήμασταν και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.